Uh, για τις αποφάσεις των συντονιστών, οι οποίες σήμερα το πρωί ήταν οι εξής. Καταρχάς, ο κύριος Χρυσόγονο θα είναι εισηγητή ε, για τη γνωμοδότηση στην ΕΚΟΝ ε, για την προληπτική εποπτεία των επενδυτικών εταιριών, όπως επίσης και για τη γνωμοδότηση στην ΕΜΠΛ για διαφανείς ε, προβλέψιμε συνθήκε εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, οι συντονιστές αποφάσισαν ε, να μην γνωμοδοτήσουν ε, επί των υπολείπων θεμάτων ε, που είχαν παραπεμφθεί στην Επιτροπή μας. Τρίτον, οι συντονιστές αποφάσισαν να μην ζητήσουν από την νομική, γνωμοδο... Ε, υπηρεσία να γνωμοδοτήσει ε, σε σχέση με αυτά που ζήτησαν οι πράσινοι για την γλυφοσάτη και συνεπώς να μην αναλυφθεί δράση ε, για το συγκεκριμένο θέμα. Τέταρτον, να εγκριθεί υποβληθούν οι προτάσεις για, τα, για το 2018, για το ερευνητικό πρόγραμμα του 2018, όπως επίσης και για την ε, αναθεώρηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος του 2017. Επίσης, το πακέτο για την πνευματική ε, ε, ιδιοκτησία να παρουσιαστεί σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Έκτον, να υποβάλουμε μία πρόταση ώστε να συμπεριληφθεί στο ελεγκτικό συνέδριο στο πλαίσιο του προγράμματος 2019 είναι μια ειδική έκθεση για την βιωσιμότητα ε, της, ε, του διοικητικού πλαισίου του Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βάσει του ψηφίσματος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9 η Ιουνίου του 2016 που αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Σημείο 7. Η δυνατότητα υποβολής από την Επιτροπή μας προφορικής ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόταση για την παράταση του πεδίου εφαρμογής για τις καταχωρισμένες σχέσεις συμβίωσης, ε, κανονισμός Βρυξέλλες 2α και κατά πόσο θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στην, συνεδρίαση της, ε, την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας ως ε, σημείο προς απόφαση. Έκτον, υποβολή προφορικής ερώτησης προς το Συμβούλιο για την πρόταση για τις, ε, για τις δημόσιες ε, εκθέσεις ε, παρακολούθησης αναχώρα για τον φόρο εισοδήματος των εταιριών για, και, να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή ΕΚΟΝ για το θέμα αυτό. Και τέλος, οι συντονιστές αποφάσισαν το προτινόμενο πρόγραμμα Κροάσεων για την κατάσταση της συλλογικής αποζημίωσης που θα γίνει το Φεβρουάριο Φεβρουάριο στην Επιτροπή μας. Αυτά λοιπόν ε, αποφασίσαμε σήμερα το πρωί με τους συντονιστές και συνεχίζουμε με τα, ζητήματα, με τα θέματα 17-18 της ημερήσιας διάταξης, την εξέταση τροπολογιών δηλαδή, για τον ε, κανονισμό περί εισαγωγής ε, της ηλεκτρονικής κάρτας ευρωπαϊκών υπηρεσιών και των ε, σχετικών, των συναφών διοικητικών διευκολύνσεων. Δεν, όμως, δεν είναι όμως εδώ η εισηγήτρια. Οπότε Oh, Μόλι ήρθε η κυρία Χάουταλα πάνω στην ώρα, γιατί δεν είναι εδώ οι άλλοι εισηγητές, οπότε τώρα θα συζητήσουμε το θέμα 19 που αφορά την εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και την ε, ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Χαούταλα, έχετε το λόγο. Δώστε μου ένα λεπτό μόνο, εφόσον άλλαξε η σειρά εξέταση των θεμάτων, να πάρω τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, μιλούμε για μια γνωμοδότηση που αφορά τον πλουραλισμό και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς ε, είναι ε, κάτι το οποίο πολλές φορές ανακύπτει συχνά μετά στις, ε, ως τμήμα του πολιτικού θεματολογίου των οργάνων μας, γιατί η ελευθερία και ο πλουραλισμός ε, των μέσων ενημέρωση δεν είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ποτέ δεδομένο και υπάρχουν ε, πολλά ε, προβλήματα ε, στα κράτη-μέλη, σε πολλά κράτη-μέλη, γιατί υπάρχει έλλειψη ε, σωστής εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού όσον αφορά την πρόληψη της κατάχρησης θέσης, δεσπόζουσας θέσης κάποιων μέσων ενημέρωσης σε διάφορες χώρες. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να θίξω αφορά ε, το να εξεταστεί επιτέλους ε, η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης και ε, το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θέσω στο πλαίσιο της γνωμοδότησης αυτής είναι κάποια νομοθετικά και διοικητικά μέτρα τα οποία χρησιμοποιούνται σε κάποια κράτη-μέλη για να, περιοριστεί και, να περιοριστούν και να ελέγχονται τα μέσα ενημέρωσης άμεσα ή έμεσα ε, γι' αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω την θεμελιώδη σημασία της ε, ε, ανεξαρτησίας των σύντακτων από πολιτικά συμφέροντα και πρέπει να πούμε επίσης ότι πρέπει να είναι δίκαιη, αμερόληπτη και διαφανής η κάλυψη των προεκλογικών περιόδων. Κάτι ακόμη, ένα ακόμη στοιχείο είναι η δυσφήμιση ε, θα θυμάστε ότι υπήρξαν συστάσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από άλλους φορείς ότι η δυσφήμιση δεν θα έπρεπε να ε, διέπεται από την ποινική δικαιοσύνη αλλά από τον αστικό κώδικα. Οπότε προτείνω να ε, ζητήσουμε να εξασφαλιστεί ότι η δυσφήμιση ε, αποποινικοποιείται και πλέον ε, θα εξετάζεται σε επίπεδο αστικού δικαίου σύμφωνα με ε, τα, τις προδιαγραφές τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς. Κάτι ακόμη ε, το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ είναι η σημασία των καταγγελόντων ε, ως βασική πηγή διερευνητικής δημοσιογραφίας. Οπότε προτείνω να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει ε, προστασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους καταγγέλλοντες, στο πλαίσιο της δημοκρατίας και της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης. Πέμπτο σημείο, η καταπολέμηση καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων ε, ε, είναι ε, μια παραπλάνηση η οποία εσκεμένα γίνεται από κάποια μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν θα έπρεπε να περιορίζει την ελευθερία ε, των μέσων ε, πρέπει απλώς ε, να δοθούν απαραίτητοι πόροι για την αντιμετώπιση αυτής της παραπλάνησης και των ψευδών ειδήσεων και πρέπει να αναγνωρίσουμε των, των μέτρων της Task Force επί του θέματος αυτού και η δημιουργή, της δημιουργικής μιας ομάδας υψηλού επίπεδου για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπλανητικής πληροφόρησης το σχέδιο γνωμοδότησης ε, είναι πάρα πολύ ε, περιορισμένο ε, ως προς το μήκος του. Αυτοί είναι οι κανόνες. Εγώ ως εισηγήτρια, όπως κάνω συνήθως, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι σε αυτήν την γνωμοδότηση. Είναι μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών ε, αυτό θα ήθελα να ε, το υπενθυμίσω. Κύριε Ρόντε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Χάουτελα για την δουλειά της. Εγώ υποστηρίζω την πρόθεση της κυρίας Χάουτελα, ωστόσο θα ήθελα να σκεφτείτε ε, το εξής, να φανταστείτε το εξής. Ε, οι αρχιδιστά, τις, ε, οι αρχισυντάκτες της ρωσικής ραδιοτηλεόρασης, εγώ λέγομαι Χένσεν, είμαι υπεύθυνο ασφαλείας του Υπουργείου Εξωτερικών της Σουηδίας και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι 600 ε, υποβρύχια ε, και F-16 θα πάνε τα μεν ε, στην, στον εύξηνο πόντο και τα άλλα στην Συρία. θα ήθελα να σας πω επίσης ότι οι ευρωβουλευτές οι περισσότεροι είναι παιδεραστές και υπάρχουν μάλιστα και πάρα πολλοί κατάσκοποι οι οποίοι έχουν σκοτώσει πάρα πολλούς ανθρώπους στις Βρυξέλλες. Χαίρομαι που γελάτε γιατί αυτές οι δύο ιστορίες που μόλις σας είναι προφανώς ψευδείς ειδήσει ε, και ε, ε, ψέματα αν όμως ήμουν επικεφαλής ασφαλείας ε, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδία και έγραφα τόσο απαράδεκτα και άσχημα πράγματα ε, σε όχι πολύ ε, φιλικά, όχι τόσο, τόσο φιλικά και δημοφιλή μέσα, τι θα έπρεπε να κάνω, θα έπρεπε να κυκλοφορώ ελεύθερος, θα έπρεπε και εγώ δηλαδή να προστατεύομαι σύμφωνα με αυτά που λέει η κυρία αλλά Το ερώτημά μου λοιπόν είναι ποια είναι η αποψή σα γι' αυτό. Ξέρω ότι ακούγεται εντελώ τρελό γιατί ποιο θα τα έκανε αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια όμω είναι ότι κανεί δεν ξέρει ποτέ και τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Εγώ δουλεύω στα μέσα μαζική ενημέρωση από το 1994 και να σα πω την αλήθεια, πιστέψτε με, κάποιοι άνθρωποι θα πούν οτιδήποτε για να ε, συκοφαντήσουν ή να δυσφημίσουν, να φέρουν σε δύσκολη θέση κάποιον. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να δούμε δούμε την πολιτική πίεση που υπάρχει κατά κάποιων ε, μέσων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να το συγχαίουμε με υποστήριξη στους καταγγέλλοντες και με το να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να αποσύρουν νόμους οι οποίοι εξασφαλίζουν ε, το προσωπικό σου νομικό δικαίωμα, νόμικο δικαίωμα προστα... προστασίας από δυσφήμιση που δεν, μέσω στοιχείων που δεν μπορούν να αποδειχθούν. Αν λοιπόν γίνει, υπάρξει αυτή η προστασία για τους καταγγέλλοντες, θα έπρεπε να υπάρχει νομίζω μία κάπως πιο μέτρια διατύπωση στα σημεία 3-4 ε, πριν οι φιλελεύθεροι τα υποστηρίξουν. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω μία σαφή διάκριση μεταξύ ε, των κατηγοριών και των προσβολών. Δεν θα έπρεπε να αποποινικοποιηθεί για παράδειγμα το να λέμε, να κατηγορούμε την κυρία Χάουταλα ε, ότι είναι κατάσκοπος. Ε, πράσινη συνεχώ συνεχώς ε, κατηγορούν τους συναδέλφους ε, ε, ε, τους συναδέλφους της δεξιάς όταν διαφωνούν μαζί τους. Όσον αφορά τους καταγγέλλοντες, εγώ συμφωνώ ότι μπορεί να αποτελεί μια πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών, αλλά θα μπορούσε να είναι και το ακριβές αντίθετο. Οπότε... Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι εμείς φυσικά υποστηρίζουμε την πρόθεση της γνωμοδότησης ε, της κυρίας Χάουτελ, απλώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να την εξισορροπήσουμε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι κάποιος θα κόψει τις προτάσεις που είπατε για την κυρία Χάουταλα και όπως επίσης το Sputnik και άλλες, τέτοιους, άλλες τέτοιε, τέτοιου είδους λέξεις. Ε, ε, φαντάζομαι ότι αυτά τα νέα θα φτάσουν στο ευρύ κοινό. Κυρία Ρέγνερ. Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για μια εξαιρετική αν και απαραίτητα σύντομη ε, γνωμοδότηση και επειδή είναι ακριβώς σύντομη είναι έξυπνη κίνηση να δούμε αν, πού μπορούμε να δώσουμε την προσθέμενη αξία στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Και πρέπει να πω ότι η προστασία των καταγγελτών είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει με πολλές λεπτομέρειες και έκθεση της κυρίας Ζωζιέ που ήταν εξαιρετική και που έγινε νομίζω και μάλλον υποστηρίχθηκε από πολλές πολιτικές ομάδες καθώς και το σχέδιο οδηγίες που πρότειναν οι πράσινοι ως τρόπο αντιμετώπισης ε, νομίζω πως μας βοήθησαν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αναφέρθηκαν. Δεν σημαίνει η προστασία του καταγγέλτη ότι σου επιτρέπεται να κάνεις ε, ψευδείς καταγγελίες και, να, ε, και κατηγορίες. Αυτά όλα γίνονται υπό την ε, πίστη ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αληθινές κάθε φορά, αλλά όχι ότι οποιοδήποτε δήλωση ό,τι κατεβεί του καθενός δηλαδή θα προστατεύεται. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει διαφοροποίηση και νομίζω ότι το να φέρουμε στην χρηματοδότησή μας είναι πολύ καλή ιδέα. Ήδη ανέφερα ότι απαραίτητα το κείμενο είναι, αναγκαστικά μάλλον το κείμενο είναι σύντομο και αν έπρεπε να, αν είχα μια ευχή εγώ αυτό θα, που θα ήθελα να προσθεθεί είναι ότι εφόσον είμαστε επίσης αρμόδιοι για τα θέματα της χρηστής ε, διοίκησης, διαχείρισης, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς έχει χρησιμοποιηθεί η νομοθεσία περί ελεύθερης πληροφόρησης ε, και τους τελευταίους μήνες θα πρέπει να δούμε ότι όταν πρόκειται ε, για τον κανονισμό 149 του 2001, δηλαδή ελεύθερη έκφραση, η Επιτροπή ή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα βλέπουμε ότι κάποιες φορές οι δημοσιογράφοι έχουν πάρει απαντήσεις που εγώ πιστεύω δεν είναι σύμμορφες με τον κανονισμό. Δηλαδή η ελευθερία ενημέρωσης έχει ε, απορριφθεί αλλά επί ε, ασταθούς ε, βάσεις και συχνά οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί δεν έχουν τα χρήματα που χρειάζονται για να τρέχουν στα δικαστήρια ώστε να απαιτήσουν τις πληροφορίες αυτές οπότε ως ε, κοινοβούλιο έχουμε ευθύνη να θυμίσουμε στην Κομισιόν και σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα Ποιε είναι οι υποχρεώσεις τους σύμφωνα με αυτό το κανονισμό και να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για το βελτιώσουμε αν πρέπει να το ξανανοίξουμε, αν πρέπει να υπάρξουν προσθήκες η επιλογή των θεμάτων είναι πολύ καλή ψευδής είναι ένα μοντέρνος, μια μόδα, είναι ένα νέο όρο, δεν είναι όμως νέο το φαινόμενο και είναι χρήσιμο να καλυφθεί, αλλά δεν θα πρέπει να αποτελεί το μόνο θέμα που μας απασχολεί στην γνωμοδότησή μας, γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί τομείς όπου πιστεύω ότι εμείς με τις αρμοδιότητές μας, ε, όπως ας πούμε για την προστασία των καταγγελτών και την προστασία Τις ενημέρωσης μπορούμε να συμβάλλουμε στην εργασία που ήδη γίνεται, στην προσπάθεια που ήδη γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Σβιεύκα. E, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ενδιαφέρον είναι αυτό το θέμα και σίγουρα θα μπορούσε κανείς να γράψει και πολλά περισσότερα σε μια μακριά έκθεση και όχι μόνο κάτι τόσο, μια τόσο σύντομη έκθεση και συμφωνώ με τα όσα είπε η συνάδελφος στην υπεράσπιση, για την υπεράσπιση δε των ε, καταγγελτών Συμφωνώ ότι πρέπει να δίνονται οι πληροφορίες και δεν είναι όμως αυτό το πιο σημαντικό. Αυτό το θέμα του πλουραλισμού και της ελευθερίας των ΜΜΕ θα έπρεπε να είναι ο κανόνας, ο κανόνας για τα μέσα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κάπως απελπιστική κατάσταση διότι ε, αυτό συμβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι έχουμε ξεχάσει έναν από τους βασικούς κανόνες, δηλαδή τους, την ευθύνη που φέρουν για τα όσα λένε. Αν στραφούμε στους ε, κώδικες ε, διοντολογίας ε, των, της δημοσιογραφίας θα δούμε θα θυμηθούμε διάφορα πράγματα. Βέβαια, ιδανικός κόσμος δεν υπάρχει, ε, και κυρίως για τα ΜΜΕ, ε, αλλά εάν στρεφόμασταν στο κώδικα διοντολογίας, τα υπόλοιπα προβλήματα θα λύνονταν πολύ πιο απλά. Και επανέρχομαι στα όσα είπατε όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αλλά στη συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στο να αγγιηθούμε τον πλουραλισμό, ε, για τα μέσα και στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα χωρίς να φτιάξουμε άκαμπτα στεγανά. Να θυμίσουμε μόνο ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τη λέξη ευθύνη. Ευθύνη, υπευθυνότητα που είναι ε, η σημαντικότερη λέξη εδώ γιατί είναι εύκολο να καταστρέψει κανείς ένα αγαθό που κανείς ε, φτιάχνει για χρόνια ε, με ανόητα ή ψευδή άρθρα. Και μετά αν ε, το δικαστήριο πει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος, όμως η ζωή του ήδη θα έχει καταστραφεί. Αν λοιπόν αυτό το project Μάλλον, συγγνώμη, αυτό το project περιλαμβάνει πολλά καλά στοιχεία, αλλά εγώ θα εστίαζα την προσοχή στο θέμα της ευθύνης τώρα να αποφασίσουμε ότι η δυσφήμιση είναι τόσο σημαντική ε, που και αν εμπίπτει στο αστικό δίκαιο ή στο ποινικό δίκαιο και εδώ όμως πάλι το ίδιο ε, θέμα μας απασχολεί δηλαδή η ευθύνη, ποιος φέρει την ευθύνη εγώ στο παρελθόν έχω εργαστεί ως δημοσιογράφος και κάθε πληροφορία που δημοσιευόταν έπρεπε να επαληθεύεται και δύο και τρεις φορές σήμερα όμως δεν επαληθεύει κανείς τίποτα Μόλις κάτι μαθαίνει το διαδίδει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα στα ΜΜΕ τη σήμερα ημέρα. Το πρόβλημα είναι λοιπόν πολύ πιο περίπλοκο. Ευχαριστώ. Δεν είναι μόνο η προστασία των καταγγελτών. Ευχαριστώ. Όταν έχουμε να κάνουμε με το θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και με την ελευθερία αυτών, μιλάμε για θέματα που βρίσκονται στην καρδιά όλων των αξιών που μας είναι προσφυλής ως Ευρωπαίων. Για μένα η, ελευθερία, η ελευθεροτυπία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταυτότητά μας και με την ελευθερία έκφρασης. Εκτιμώ τα σχόλια που έγιναν για την ευθύνη του δημοσιογράφου και για τον έλεγχο των πηγών του. Αλλά αυτό πρέπει να συμβεί και στο πλαίσιο της δίκαιης και κατάλληλης προστασίας. Στον τομέα αυτό, οι πληροφοριοδότες είναι πολύ κρίσιμη πηγή πληροφοριών και αν εξετάσουμε τις πηγές των δημοσιογράφων εν γέννη ε, και το τι έχει να πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε διάφορες περιστάσεις, ε, βλέπουμε ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αποσιωπούνται οι πληροφορίες και βεβαίως στη Μάλτα είχαμε την δολοφονία της ε, Δάφνης Καρουάνα Γαλίσια που ήταν το πιο η πιο ακραία υπόθεση, αλλά εκεί που εμποδίζονται λοιπόν οι δημοσιογράφοι να κάνουν τη δουλειά τους ή μπας περιπτώσει δεν προστατεύονται καταλήλως, εκεί αυτό έχει ένα εφέ ε, αποτροπ, Αυτό όχι γιατί σταματάνε οι, δημοσιογράφοι, αλλά γιατί η κοινωνία χάνει αυτό το επίπεδο πληροφορίας το οποίο μπορεί να έχει μέσω των πληροφοριοδοτών ή των δημοσιογράφων που κάνουν έρευνα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ας πούμε στη Μάλτα ένας καταγγέλτης που αποκαλύπτει πράγματα που είναι ευνοϊκά για την κυβέρνηση παίρνει συμβάσεις απασχόλησης και γίνεται ε, πάμπλουτος. Άμα όμως αποκαλύψει στοιχεία για την ιδιωτική ζωή της Πρωθυπουργού, ε, ε, δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση που πρέπει να φύγει από τη χώρα. Και τώρα Καθώς έχουμε, την όπως είδατε και η αντιπροσωπεία των Ευρωβουλευτών μόνοι σας, έχουμε έναν ε, πληροφοριδότη που ονομάζεται Jonathan Fares, που θέλει να αποκαλύψει πολύ σημαντικές πληροφορίες, αλλά που επειδή δεν έχει ακόμα λάβει την προστασία του που αξίζει τον πληροφοριδότη, δεν μπορεί να αποκαλύψει τίποτα, μπορεί να εκτεθεί σε φυλάκιση ή σε ε, σοβαρά πρόστιμα. Οπότε, όντως πρέπει να προστατευτούν ε, οι πληροφοριοδότες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα. Κάτι ακόμα που, δεν, που θέλω να θίξω εδώ είναι το θέμα της εγγύησης της ελευθερίας των δημοσιογράφων και της προστασίας τους από την φήμωση. Και αυτό συμβαίνει στη Μάλτα από ε, οντότητε όπω η φυλάτο. δεν το κάνω στη Μάλτα αλλά πάνε στη ΣΥΠΑ γιατί λένε ότι υπάρχει σύνδεση από το ίντερνετ, από το facebook, από την ε, καταγραφή του ιστότοπου και τι κάνουνε τους ε, διώκουν ε, δικαστικά σε μια δικαιοδοσία που δεν έχει καμία σχέση με το πού έχουν αποκαλυφθεί οι πληροφορίες, ώστε ακριβώς οι δημοσιογράφοι να βρεθούν σε μια κατάσταση όπου να αρχίσουν να κάνουν πίσω στις πληροφορίες που δίνουν στο κοινό. Ε, άρα λοιπόν ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να προστατεύσουμε τους, με, τους, με, τους με, ε, δημοσιογράφους μας από αυτές τις διατλαντικές επιθέσεις ε, που χρησιμοποιούν την Αμερική για να φημώσουν δημοσιογράφους στις χώρες μας. Ευθύνη λοιπόν βεβαίως συμφωνώ ναι, ε, εναντίον στις παιδείς ε, ειδήσει, αλλά πάντοτε υπέρ της υποστήριξης των δημοσιογράφων και υπέρ της υποστήριξης μιας από τις πιο θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Χάουταλα που έχει συντάξει την έκθεση γνωμοδότησης και τονίζει τα πλέον σημαντικά θέματα. Δεν θα επανέλθω στην ανάγκη προστασίας των καταγγελτών. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Των καταγγελόντων, αν θέλετε. Και το γεγονό ότι σε διάφορες χώρες, όπως και, στη, και στην Γαλλία, έχουν προχωρήσει πολύ νομοθετικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, έχω δύο άλλα ζητήματα, που ίσως είναι πιο ανησυχητικά. Το πρώτο, για το οποίο μιλεί η κυρία Χάουταλα, είναι τη συγκέντρωση, σε λίγα χέρια δηλαδή, των μέσων ενημέρωσης, ε, που αντιστρατεύεται την πολυφωνία των μέσων έχω μπροστά μου μια σύνοψη βιβλίου που λέει «Οι νέες αυτοκρατορίες των μέσων» εκδοθέν προέτους και που λέει ότι 8 δισεκατομμυρίουχοι στη Γαλλία κατέχουν σχεδόν το 100% των μετοχών των ε, μεγάλων μέσων μασικής ε, ενημέρωση στην Γαλλία και μπορούν να ασκήσουν άμεση επιρροή, διότι είναι ιδιοκτήτες ή και μέσω απειλών, ότι δηλαδή θα τους κόψουν τα έσοδα από τις διαφημίσεις. Ένα παράδειγμα. Μαρτυρία δημοσιογράφου της Le Monde που λέει ότι είχε το λάθος να γράψει ένα άρθρο για το λιμάνι του Αμπιτζάν ο οποίος του επέβαλε μπλοκ στις διαφημίσεις για το έντυπό του. Επομένως η ελευθεροτυπία και η ελευθερία ε, ε, εντύπων όπως ε, εγκρήτων εφημερίδων όπως η Μοντ τελικώς δεν είναι καθόλου διασφαλισμένη. Αυτό είναι θεωρώ το μείζον πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα που επισημαίνει η κυρία Χάουταλα και την ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό είναι που επισημαίνει ότι ο αγώνας κατά των ψευδών ειδήσεων, fake news, δεν θα πρέπει να οδηγήσει τα κράτη να ε, δημιουργήσουν ένα είδος κονφορμισμού, ε, απόλυτης, ε, απόλυτου συμβιβασμού. Αυτό που χρειάζεται είναι να διαψεύδονται οι ψευδείς ειδήσει και να εξηγείται με λογικό τρόπο ότι πρόκειται για ψευδείς ειδήσει. Εγώ θεωρώ ότι έχει μυαλό ο κόσμος και θα καταλάβει πού βρίσκεται η αλήθεια. Διότι αλλιώς θα φτάσουμε σε έναν άνωθεν κομφορμισμό ή σε έναν που θα επιβάλλεται από ιδιωτικές επιχειρήσεις που ε, έχουν στα χέρια τους ε, το facebook, το ε, διαδίκτυο και το καθεξής. Και τελικώς αυτές θα ρυθμίζουν και αυτό θα ήταν το χειρότερο απ' όλα. Θεωρώ λοιπόν ότι η κυρία Χάουταλα μεγάλη υπηρεσία μας προσφέρει επισημένοντας τους δύο αυτούς κινδύνους που μας ανησυχούν για την ώρα, δηλαδή επί του παρόντος. Ευχαριστώ. Η δική σας ήταν η τελευταία παρέμβαση. Θα προσθέσω μόνο, λέει ο πρόεδρος ότι έχω συμμετάσχει σε διάφορες ε, διασκέψεις για θέματα ψευδών ειδήσεων, όπου εμπειρογνώμονες ασφαλείας έλαβαν το λόγο για να εξηγήσουν ότι η δυνατότητα αντιμετώπισης των ψευδών ειδήσεων με εξηγήσεις, με παροχή εξηγήσεων δηλαδή, θεωρούν τα πρόσωπα αυτά οι δήμονες δηλαδή ότι αυτό δεν είναι ο σωστός τρόπος. Ότι είναι εξαιρετικά ασθενη η αντίδραση αυτή. Αυτά λένε οι εμπειρογνώμονες. Τόσο πολλές πάντων το συζητούμε. Is set τροπολογίες μέχρι τις 30 ε, Ιανουαρίου. Οπότε παρακαλώ να το λάβετε αυτό υπόψη, κυρία Χάουταλα. Ναι, εγώ ως συντάκτρια γνωμοδότησης νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Αυτή η περίεργη ανταλλαγή απόψεων ήταν ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί νομίζω ότι όλοι μιλήσατε για κάτι ε, του, από το οποίο έχετε κι εσείς η ίδια εμπειρία υπό το ένα ή το άλλο πρίσμα ε, με έχουν ε, μάλιστα αποκαλέσει διπλή κατάσκοπο ένας από τους συναδέλφους σας εδώ στο κοινοβούλιο και είμαι και στη μαύρη λίστα των Ρώσων ή είμαι Ρώσα, Ρώσος κατάσκοπος, ε, Ρωσίδα κατάσκοπος είμαι διπλή κατάσκοπος εν πάση περιπτώσει ε, προφανώς πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ αυτού που θα λέγαμε ε, δυσφημιστική προσβολή τέλος πάντων ε, προσβολή και όχι κατηγορία μια ψευδή κατηγορία και ο κύριος Βεύμα νομίζω θα με διορθώσει αν κάνω λάθος, ε, πάντοτε θα αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο μιας ε, ποινική δικαιοσύνης. Προφανώς ε, θα συμβαίνει αυτό σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω όμως ότι θα έπρεπε πράγματι να δούμε τις συστάσεις κάποιων ε, διεθνών ε, ομάδων ε, επίβλεψης που μας λένε ότι το θέμα της δυσφήμισης είναι επίσης σημαντικό. Νομίζω ότι η κυρία Ρέντα μας έδωσε μια πάρα πολύ, πολύ καλή εξήγηση για ποιο λόγο η προστασία των καταγγελόντων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντική και επίσης ε, υπόθηκε ότι πρέπει να ισχύει και να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Με χαρά να ακούσω και τις δικές σας τροπολογίες. Κύριε Σβίφκα, ναι, νομίζω ότι η ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική και όταν αρχίσατε την παρέμβασή σας είπατε ότι πρέπει να πάμε στις στις... πίσω στις ε, αρχικές ε, αρχές της δημοσιογραφίας και να επενθυμίσουμε κιόλα τη σημασία της αυτορύθμισης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και αυτό είναι σημαντικό αλλά επειδή αλλάζει το περιβάλλον των μέσων μαζικής ενημέρωσης με τα ηλεκτρονικά μέσα, με το διαδίκτυο που κερδίζει έδαφος πάρα πολύ γρήγορα. Ε, όταν διαβάζω το The Guardian για παράδειγμα, κάθε φορά νιώθω ε, ένοχη όταν ε, δεν κάνω κλικ για να ε, επενέσω ας πούμε την, ε, το πολύ καλό άρθρο γιατί κάθε φορά που διαβάζει κανείς ένα άρθρο στο τέλος λέει ότι μπορεί κάποιος να κάνει μία μικρή δωρεά για να υποστηρίξει τη σοβαρή ε, δημοσιογραφία. Το ζήτημα λοιπόν των πηγών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πρόσβαση στις πληροφορίες και αυτό είναι σημαντικό. Η δημόσια πρόσβαση πληροφορίες, ο κανονισμός μας 1049-2001 για την δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα είναι ένα βασικό ε, είναι μια βασική ε, ε, νομοθετική πράξη που αφορά τη δημοσιογραφία. Κύριε Ζαμέτη, είπατε κάτι για τις στρατηγικές επιθέσεις στους δημοσιογράφους. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτι τέτοιο προς την, τον, την παρεμπόδιση μιας δημοσίευσης κάποιου είδους ας πούμε AUTHORWAVE απεριορισμού ε, μέσω απειλών ε, και να μην σας πω ότι πάρα πολλές φορές ε, συμμετέχουν και δικηγόροι επιφανείς από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όσον αφορά το θέμα των ψευδών ειδήσεων και αυτό χρήζει ιδιαίτερη προσοχή, η Επιτροπή Λίμπε και αυτή θα το εξετάζει, γιατί υπήρξαν παραδείγματα για το πού θα μπορούσε να μας οδηγήσει κάτι τέτοιο και υπάρχει επίσης και ένας για τη δημόσια ασφάλεια, γιατί εξ όσων είναι πάρα πολύ εύκολο να φυτέψει κανεί με πολύ στρατηγικό στόχο ψευδείς ειδήσει για να δημιουργήσει διεθνεί συγκρούσει. Νομίζω ότι η κατάσταση λοιπόν με το Κατάρ ε, ε, πριν από λίγο καιρό μπορεί να, αποτε... να ήταν αποτέλεσμα ε, τέτοιου είδους εμφύτευσης ψευδών ειδήσεων σε κάποιο πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ θα αντιμετωπίζουμε πολύ συχνότερα τέτοιου είδους περιπτώσεις όταν υλικό ειδήσεων ή οπτικοακουστικό υλικό, οπτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολύ ε, ψευδή τρόπο ώστε να δοθεί μία ε, ψευδής εντύπωση για το τι συμβαίνει στην άλλη άκρη του κόσμου και επί του οποίου κανείς δεν έχει έλεγχο στην πραγματικότητα για να μπορέσει να ελέγξει κανείς την άποψη κοινή γνώμη. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Χάρηκα πολύ με αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Θα περιμένω στις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Αυτά για αυτό το σημείο. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τα ε, σημεία 17 και 18. Εξέταση τροπολογιών για τον κανονισμό περί εισαγωγής μιας ηλεκτρονικής κάρτας ευρωπαϊκών υπηρεσιών και των ε, σχετικών οδηγιών. Η κυρία Γκέπχαρτ έχει το λόγο που είναι η συγγήτρια για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω πολλά να σας εξηγήσω. Δηλαδή περισσότερα από τα όσα είχα αναπτύξει την προηγούμενη φορά που έκανα την πρόταση, μάλλον δύο προτάσεις. Είπα δηλαδή να παραπεμφθούν εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει ξανά κείμενα πιο συνεκτικά και με πιο ανάγλυφες τις λεπτομέρειες της διασυνδέσεως των διαφόρων μηχανισμών που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των μηχανισμών της ε, υπηρεσίας και την παροχή υπηρεσιών, καθώς και, και για την αμοιβή αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή και αυτά που προετοιμάζουμε τώρα σε σχέση με την ψηφιακή πύλη. Γιατί αυτό θα πρέπει να είναι τελικό και η προστιθέμενη αξία των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό είπα και εγώ, α παραπενθούν εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επομένω δεν έχω καταθέσει τροπολογίε, διότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν και συνεπέ. Αναμένω με ενδιαφέρον τώρα τι θα πούν οι συνάδελφοί μου που έχουν υποβάλει τροπολογίες. Ο Ράγεφ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Ο κύριος Μπούντα είναι κολλιόμενος σήμερα και θα διαβάσω εγώ κάτι που μου έχει δώσει για το συγκεκριμένο θέμα. Λέει ο κ. Μπούντα ότι θα ήθελε πρώτα να τονίσει ότι είναι αντίθετος με την παραπομπή εκ νέου του ε, σχεδίου οδηγίας και κανονισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι θα ήθελε να βελτιώσει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πρωτολογίες τις οποίες καταθέτει ον πεπισμένος ότι έχουν χρησιμότητα και ότι θα μειώσουν τη γραφειοκρατική επιβάρυνση στους παρόχους υπηρεσιών που επιθυμούν να παράσχουν υπηρεσίες διαμεθοριακά. Στη βάση των νέων λοιπόν μηχανισμών που ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούν να γνωρίζουν τι πρέπει να αναμένουν από τις διάφορες εθνικές αρχές. Με τις δικές μου τροπολογίες, λέει ο κύριος Μπούντα, θεωρώ ότι η αποτελεσματική χρήση της ε, κάρτας ηλεκτρονικών υπηρεσιών δεν αντιβαίνει ούτε την ουσία ούτε το πεδίο εφαρμογή τη νέα οδηγία. Άλλωστε δεν έχει σχέση ούτε με την απόσπαση εργαζομένων, δηλαδή με τη σχετική οδηγία, ούτε επηρεάζει τους υφιστάμενους κανονισμούς, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού για την παροχή υπηρεσιών, όπως κοινωνική προστασία, προστασία καταναλωτών, υγεία και ασφάλεια ή περιβάλλον. Για αυτούς τους λόγου συνεχίζει ο κ. Μπούντα, καταθέτω, λέει ο ίδιο, δηλαδή, ως κατευθυντήρια αρχή την αρχή της χώρας προελεύσεως. Για την ηλεκτρονική κάρτα λέει υποβάλλω τροπολογίες για να διευκρινίσω πώς μπορεί να εφαρμοστεί η ιδέα αυτή τονίζοντας και πάλι την εθελοντική φύση του μηχανισμού. Σε ό,τι αφορά το στοιχείο του κόστους, θεωρεί ο κύριος Μπούντα ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις για την Ένωση θα είναι μάλλον μετριοπαθείς και επιπροσθέτως τονίζει ότι η κεντρική διαχείριση των ηλεκτρονικών καρτών θα πρέπει να είναι δωρεάν η υπηρεσία την οποία θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε ό,τι αφορά το κόστος σε βάρος των παρόχων υπηρεσιών, αυτό θα μειωθεί σημαντικά, δοθέντος του ότι η σχετική τεκμηρίωση θα απαιτείται μόνο άπαξ. Θεωρώ λοιπόν ότι η βελτιώσεις που προτείνω, λέει πάντα ο κ. Μπούντα, θα επιτρέψουν στους παρόχους υπηρεσιών στη βάση της ηλεκτρονικής κάρτας να ξεπεράσουν την αβεβαιότητα του νομικού περιβάλλοντος σε διάφορες χώρες μέλη, την ανάγκη να συμπληρώνουν έντυπα σε διάφορες γλώσσες, την ανάγκη να μεταφράζουν τα εγγραφά αυτά, να ε, βεβαιώνουν τη γνησιότητα των εγγράφων. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούν έτσι να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών τους και να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες εν τέλει. Ευχαριστώ. Ζλωτόφσκι. Ευχαριστώ, φίλε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Και στο όνομα της ομάδας μου ECR θα σας πω ότι η θέση μας είναι ότι η πρόταση της Κομισιόν παρά τις κάποιες ελλείψεις είναι χρήσιμη. Δεν συμφωνώ με, με τις τροπολογίες που ζητούν απόρριψη της προτάσεως. Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να τροποποιηθεί η πρόταση της Κομισιόν έτσι ώστε να είναι πιο ευεφάρμοστη και να διευκολύνει τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε διαμεθοριακό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Κάρτα, η CARD, δεν θα χρησιμοποιηθεί για να καταστρατηγήσει εθνικούς μηχανισμούς, αλλά θα μας επιτρέψει να δράσουμε αποτελεσματικά και απέναντι σε ξένες εταιρείε. Στην τροπολογία 13 λέτε ότι αυτό δεν θα αλλάξει τις αρχές της απόσπασης εργαζομένων, γιατί το θέμα αυτό είναι ε, ιδιαίτερα ευαίσθητο. Θα είναι οικειοθελής ο μηχανισμός αυτός. Σωστό. Οι τροπολογίες του, της ομάδας ECR στοχεύουν στη ρύθμιση κάποιων λεπτομεριών. όπως των επαληθεύσιμων λεπτομεριών, καθώς και τις προθεσμίες που ισχύουν για την δημόσια διοίκηση, οι οποίες για την ώρα είναι πάρα πολύ βραχίες. Στην τροπολογία παριθμών 100 προβλέπουμε ένα μηχανισμό με τον οποίο μπορεί να εκδίδεται η ηλεκτρονική κάρτα αν και δεν θα καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις. Η δική μου έκκληση λοιπόν είναι να μην απορρίψετε το σύνολο της προτάσεως της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορούμε να είμαστε σύντομες. Συμφωνούμε με την εισηγήτρια ότι δηλαδή πρόταση υπερβαίνει κάποια όρια και δεν είναι καλά επεξεργασμένη. Δεν είναι λοιπόν σαφές για μας εάν επηρεάζεται η οδηγία παροχής υπηρεσιών, εάν πηγαίνει να βάλει την αρχή της χώρας προέλευσης από την πίσω πόρτα και η κυρία Γκέπχαρτ από την εμπειρία της με την οδηγία απόσπαση εργαζομένων μπορεί να το κρίνει αυτό καλύτερα. Θεωρούμε και εμείς λοιπόν ότι πρέπει να παραπεμφθεί εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση για να συζητήσουμε ξανά την βάση του θέματος για το πώς θα εξασφαλιστεί και θα ρυθμιστεί η ελευθερία παροχής υπηρεσιών που όμως νομίζω δεν μπορεί να γίνει με το παρόν έγγραφο της Κομισιόν. Le Breton. Moi, impression depuis έχω την εντύπωση ότι αυτή η υπόθεση δεν έχει προετοιμαστεί σωστά, γιατί η πρόταση μας υποβάλλει σήμερα η Κομισιόν έρχεται, είναι πρώιμη. Δεν έχει οριμάσει το θέμα. Και τα όσα λέει η κυρία Γκέπχαρτ με βρίσκουν σύμφωνο ε, και ειδικά εκεί που λέει ότι δεδομένων των προθεσμιών που πρέπει να τηρηθούν και ότι ε, δεν έχουμε αρκετές διευκρινήσεις, νομίζω πως εδώ έχουμε φτάσει σε απάτες, σε δημιουργίες πλαστών ε, ταυτοτήτων και νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα από αυτό που θέλουμε να λύσουμε. Είμαι υπέρ λοιπόν του να απορριφθεί ως έχει αυτό το σχέδιο και να μην ακολουθηθούν άλλες οδοί, όπως ας πούμε να ανανεωθούν οι φυστάμενες οδηγίες. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει άλλος κανείς το λόγο. Κύριε Κέπχαρτ, θέλει να προσθέσει τίποτα? Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την εργασία που έχετε καταβάλει ορισμένοι εξημών, αλλά εξετάζοντας τις τροπολογίες σας, βλέπω πολλές που ζητούν διαγραφή ολόκληρων παραγράφων της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή που κάνουν κάποια οριοθέτηση με, τους υφιστάμενους, με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις. Εκεί φαίνεται καθαρά το πρόβλημα της πρότασης αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν είναι καλοχωνεμένη ακόμα και ότι εν τέλει κάνει λιγότερα πράγματα υπέρ της, ευρω... της ενιαίας αγοράς, υπέρ ε, ε, λιγότερα μάλλον υπέρ της ε, πρόσβασης, διότι περιπλέκει τα πράγματα ακόμη περισσότερο και ιδίω για τι επιχειρήσει, ιδίω για τι μικρέ και μεσές επιχειρήσει. Θα καταστήσει το έργο του ακόμη δυσκολότερο <clears throat> να παρέχουν δηλαδή τι σχετικέ υπηρεσίε. Για μένα θα ήταν πολύ καλύτερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα ξανασκεφτεί τα πράγματα αυτά όλα από την αρχή και να φροντίσει ώστε όλες οι ρυθμίσεις που έχουμε ήδη να εφαρμοστούν στις χώρες μέλη με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν και να αποδίδουν καλά. Διότι έχουμε τον ενιαίο συνομιλητή, έχουμε την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, έχουμε το, την ψηφιακή πύλη που βρίσκεται τώρα υπό κατασκευή. Έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φοβούμε ότι αν έρθουμε τώρα να προσθέσουμε κάτι ακόμη, ε, πια οι επιχειρηματίες δεν θα ξέρουν καν που να στραφούν και πώς θα διεκδικήσουν τα δικιά τους. Θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιηθούν οι μηχανισμοί που υπάρχουν ήδη και που δεν λειτουργούν καλά. Το δέχομαι αυτό. Εκεί χρειάζονται λοιπόν βελτιώσεις. Αλλά δεν χρειάζεται νέο εργαλείο το οποίο ούτε και αυτό θα λειτουργήσει σωστά και εν τέλει θα σημάνει περισσότερες δυσκολίες για την ενιαία αγορά παρά καλό. όταν βλέπουμε ότι δημιουργούνται νέε αρχέ και μάλιστα νέα κεντρική αρχή, το οποίο βεβαίω έχει και κόστο για τι χώρε μέλη. Του δυσκολεύει τη δουλειά. Δυσκολεύει και την δουλειά των κρατών μελών δηλαδή, αντί να τη διευκολύνει. Δεν προσπαθώ να εμποδίσω την ύπαρξη και λειτουργία της ενίας αγοράς. Θέλω να απλουστευτεί, να διευκολυνθεί και να μην γίνει πιο περίπλοκη για τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ζητήσει να λάβει το λόγο. Ναι, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Να τονίσω το εξή. Η προπαρασκευή, προπαρασκευή της προτάσεως ήταν μακροχρόνια εντατική με πολλές διαβουλεύσεις. Μιλήσαμε με πολλούς ενδιαφερομένους ε, τομείς. Μιλήσαμε για τα σχετικά κολλήματα, κάθετος εμπόδια θα είναι οικειοθελής ο μηχανισμός αυτός, Εθελοντικό και καμιά επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να τον χρησιμοποιήσει παρά μόνο αν θέλει. Άρα δεν θα είναι έξτρα επιβάρυνση. Εμποδίζει την εφαρμογή της οδηγία υπηρεσιών. Όχι. Ανοίγει την ε, αρχή της χώρας προελεύσεως, την ξαναφέρνει δηλαδή από την πίσω πόρτα. Όχι, με κανένα τρόπο. Δηλαδή το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επαναλάβω ε, τα όσα έχω ήδη πει. Δηλαδή πρόκειται για μια μετριόφρονα προσπάθεια να διευκολύνει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι όλο. Okay. Ε, just let me inform you. Να σας ενημερώσω απλώς ότι η έγκριση προβλέπεται ε, στη συνεδρίασή μας 21 και 22 Φεβρουαρίου για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο και πάμε στο 20 που αφορά τις συμβάσεις για την υποβολή ψηφιακού για, στις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Θα θέλαμε πάρα πολύ, κυρία Γκέπχαρτ, να παραμείνει. Είναι μία από τους συνεισηγητέ, αν όχι τουλάχιστον ο κύριος Φως. Ευχαριστώ. Μετά από την ικανοποιητική πορεία των ψηφοφοριών στην Επιτροπή τον ε, Νοέμβριο, άρχισε ο τριμήρης διάλογος στις, ε, τον Δεκέμβριο στις 5 και στις 12 Δεκάτου Έγιναν λοιπόν δύο συνεδριάσεις τριμήρους διαλόγου. Στις 5 είχαμε συζητήσει τα άρθρα 6 και 6α για τα κριτήρια συμβατότητας ε, του συμβατικού αντικειμένου και αρχίσαμε επίσης να συζητούμε και το άρθρο 15 και τις αλλαγές του ε, ψηφιακού περιεχομένου. Στις 12 12 δεύτερη συνεδρία τριμήρους διαλόγου άρθρα 9 και 10 που αναφέρονται στην ευθύνη του πολιτού και στο βάρος αποδείξεως και άρθρο 12 για την ιεράρχηση των νομικών ε, συνεπειών. Έχουν ε, οργανωθεί άλλοι δύο τριμερείς διάλογοι, 30 πρώτου, τώρα Βουλγαρική Προεδρία πλέον, θα γίνει τρίτη συνεδρία τριμερούς διαλόγου πάλι για το άρθρο 15, δηλαδή τροποποιήσεις ε, ψηφιακού περιεχομένου και θα εξετάσουμε πάλι τα άρθρα 13 και 16 που αναφέρονται στον τερματισμό των συμβάσεων αυτών. Άλλη συνάντηση διαλόγου θα είναι για τις 6 Τρίτου. Συνολικά νομίζω η πρόοδος είναι επαρκής ε, για όλα αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν και ιδίως ό,τι αφορά την διασύνδεση μεταξύ βασικού κανονισμού προστασίας δεδομένων και συμβατικού δικαίου Εκεί θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες συνταλλαγές απόψε ακόμη, αλλά και στο πολιτικό επίπεδο και ιδίω εκεί συζητήθηκε τώρα δεδομένα ως αντιπαροχή το θέλουμε αυτό, ναι ή όχι. Μιλούμε εκεί και για την embedded software και για το επίπεδο της εναρμόνισης, για τις εγγυήσεις, για το βάρος αποδείξεως και ούτε καθεξής. Όλα αυτά τα πράγματα θα χρειαστεί να τα ρυθμίσουμε. Εν τέλει πάντως νομίζω ότι έχουμε κάνει ε, πρόοδο και μάλιστα αρκετά σημαντική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Κρίμα που είναι τόσο λίγοι συνάδελφοι παρόντες. Ειδικότερα στους συνεισηγητές αναφέρομαι. Θέλει κανένας άλλος συνάδελφος να σχολιάσει? Μάλλον όχι. We close this item, yes. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και πηγαίνουμε στο 21. Πού είναι? η παρακολούθηση κατοξιδών συμπράξεων και άλλων εφαρμοστικών μέτρων. Κύριε Λεμπροτών, είστε εισηγητή για το θέμα αυτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη φορά πρόκειται για ένα διεθνές πρότυπο, το EFRS ε, λογιστικό πρότυπο, το υπαριθμό 9, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το συγκεκριμένο πρότυπο. Βάσει του άρθρου 106 εμείς πρέπει να επαληθεύσουμε τις κατεξοδότηση πράξη, τις εκτελεστικές πράξεις, συγγνώμη. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν βλέπω καμία αντίρρηση, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αντίφαση σε σχέση με ε, την, ε, το διεθνές αυτό πρότυπο οπότε δεν έχω τίποτε περαιτέρω να πω. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ε, δεν βλέπω και άλλα σχόλια από τους συναδέλφους, άρα μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το σημείο 21. Για το 22 τώρα, για την επικουρικότητα, το σημειώνουμε και... Μία ακόμη ενημέρωση η επόμενη μας συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 21 και 22 Φεβρουαρίου. Αυτό είναι το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας για σήμερα. Οπότε κηρύσω το πέρας της συνεδρίασης.